όπου αφορά τις αλλαγές στις επιτροπές ε, και στις αντιπροσωπείες. Ο καταλόγος με τα ονόματα αυτά θα επισυναυθεί στα πρακτικά της συνόδου μας και θα θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί εάν κανείς δεν φέρει αντίρρηση, δεν προβάλλει αντίρρηση όσον αφορά αυτό τον κατάλογο. Το επόμενο σημείο της ημερησίας διαταξής μας αφορά τη δήλωση